Το λόγο έχει και πάλι ο Επίτροπος κύριος Χάν. Κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, από την αρχή της εντολής μας η βελτίωση των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική ήταν από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας. Η συνάντηση κορυφής Ένωσης ΣΕΛΑΚ είναι ένα παράδειγμα αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε, να βρούμε δηλαδή βιώσιμες λύσεις σε παγκόσμιες απειλές. Η ενίσχυση των σχέσεων με την Κούβα είναι βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της βελτίωσης των σχέσεων αυτών είναι η ταχύτητα με την οποία έγινε η βελτίωση και προσβλέπουμε και σε περισσότερες θετικές αλλαγές. Δεν πρέπει να χάσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και είναι πολλές για να μην παραμείνει η Ευρώπη ουραγός αλλά να καθοδηγεί τις εξελίξεις. Τους τελευταίους μήνες η υπάτη εκπρόσωπος ε, ήρθε σε προσωπικές επαφές με την κουβανική πλευρά και η πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντίνα έγινε με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας, Ροντρίγκε. Και ύστερα έγιναν επαφές και με τον Ραούλ Κάστρο για θέματα επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου. Μετά ο Υπουργός Εξωτερικών Ροντρίγκες ήρθε στις Βρυξέλλες για να ξαναρχίσει ένας επίσημος πολιτικός διάλογος και στα περιθώρια της διάσκεψης ε, ΣΕΛΑΚ Ένωσης έγιναν και άλλες επαφές. Το Φεβρουάριο του 2014 η Ένωση ενέκρινε οδηγία για τον πολιτικό διάλογο και, ε, συμφωνία συνεργασίας τη λεγόμενη PTCA για την Κούβα για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και Κούβας. Αυτό μετά από μακρά διαδικασία συζητήσεων στο Συμβούλιο με την καθοδήγηση του Προέδρου Κάστρο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι όντως κάνουμε προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεών μας με την Κούβα. Η ενθάρρυνση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κουβανών. Θα συμπεριλάβουμε θέματα πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Απρίλιο του 2014 και οργανώθηκαν διάφοροι γύροι τους όπως τον Αύγουστο και τον Μάρτιο του 2015. Η κυρία Μογκερίνη ήρθε σε επαφές και τους περασμένους μήνες με την κουβανέζικη πλευρά και στις 16 Ιουνίου οι διαπραγματευτές ξανασυνήλθαν στις Βρυξέλλες συζήτησαν σε επικοδομητικό κλίμα και ατμόσφαιρα και καταφέραμε σημαντική πρόοδο ιδιαίτερα για τον διάλογο για την ε, συνεργασία. Τα, επόμενα, τα υπόλοιπα κεφάλαια προχωρούν και μάλλον θα κλείσουν στον επόμενο γύρο των συζητήσεων. Για το πολιτικό θέμα επίσης υπήρξε πρόοδος, οι διαπραγματευτές έκαναν ανταλλαγή απόψεων και αποσαφινίστηκαν οι θέσεις τους έτσι ώστε να υπάρξει μια σε μεγαλύτερο βάθος προετοιμασία για τον επόμενο γύρο αρχές Σεπτεμβρίου. Ίσως γνωρίζετε ότι συμφωνήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Ροντρίγκε να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις και σύντομα να καταλήξουν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα ήταν προς αμοιβαίο τους όφελος. Η πρόοδος στο γύρο αυτό δείχνει τη δέσμευση που έχουν και οι δύο πλευρές για τη βελτίωση των σχέσεών τους. Επίσης σημειώθηκε πρόοδος σε έναν τομέα που είναι στη βάση των σχέσεών μας με την Κούβα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερίας. Το Μάρτιο προτάθηκε στον, στον Υπουργό Εξωτερικών Ροντρίγκε να γίνει ένας δομημένος διάλογος ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τον πολιτικό διάλογο στις Βρυξέλλες συμφωνήθηκαν συμφωνήθηκε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και για τον διάλογο αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρώτη του συνάντηση έγινε στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουνίου υπό την ηγεσία του Σταύρου Λαμπρινίδη με σκοπό να συμφωνηθεί η μορφή και η στόχη του διαλόγου αυτού πριν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις PTCA. Έτσι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα σχεδιαστεί με βάση την γενικότερη συμφωνία και θα μας δώσει μία ευκαιρία να βελτιώσουμε την αμοιβαία κατανόηση για ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, να γίνει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και εμπειριών και να ταυτιστούν πιθανή τομή συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και Κούβας. Επίσης, μας δίνει ένα βήμα για να συζητιούνται και με μονομένες ατομικές περιπτώσεις. Ο διάλογος αυτός λοιπόν θα χορηγήσει περισσότερη πληροφόρηση και θα συνοδέψει τον επίσημο πολιτικό διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, με βάση αυτές τις θετικές εξελίξεις, είναι απογοητευτικό αυτό που μάθαμε ότι έγινε την περασμένη Σαββατοκύριακο στη Χαβάνα δηλαδή βιαιοπραγίες. Δεν υπάρχει λόγος να περιορίσει κανείς την ειρηνική έκφραση απόψεων και να υπάρχει βία καταπίεση ειρηνικών διαδηλωτών. Η άσκηση της εξουσίας πρέπει να γίνεται με συγκράτηση. Αναμένουμε από τις κουβανικές αρχές να πάρουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να διορθωθούν αυτά. και του ζητούμε να επιτρέψουν οποιαδήποτε ειρηνική έκφραση απόψεων. Επίσης, εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας και σε θέματα εξωτερικών σχέσεων με την Κούβα όπως με την Κολομβία. Επίσης γενικότερη συνεργασία σε υγειονομικά θέματα όπου παίζει σημαντικό ρόλο η Κούβα ή συνεργασία για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών με ενόψη της σχετικής διάσκεψης των Παρισίων. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει και το θέμα του πλησιάσματος της Κούβας με τις Ηνωμένε Πολιτείες που πρόσφατα γιατί πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα, θα αρχίσουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτό συμφώνησαν ο πρόεδρος Ομπάμα και Κάστρο, οι πρόεδροι Ομπάμα και Κάστρο. Η απομόνωση της Κούβας δεν έχει πια νόημα σήμερα. Είναι απομεινάρι του ψυχρού πολέμου και θα πρέπει να λήξει. Αυτό ιδιαίτερα για μας τους Ευρωπαίους που για δεκαετίες υποφέραμε από τη διαίρεση που δημιούργησαν οι σχέσεις του ψυχρού πολέμου. Και ελπίζουμε σύντομα να λήξει και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας που είναι τελείως άχρηστο και αντιπαραγωγικό. Και έχει και αρνητικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικά στην Κούβα. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το λόγο έχει ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τις ε, πλήρεις ε, λεπτομεριακές ε, πληροφορίες γεμάτο ελπίδες που μας δώσατε. Είναι σαφές ότι ο εμπορικός διάλογος προχωρά είναι σαφές επίσης από τις εκφράσεις ε, των διπλωματών ότι ο πολιτικός ε, διάλογος ε, παραμένει στους όρους του παρελθόντος. Πιστεύω, Πρόεδρε Επίτροπε, το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία πολιτικού διαλόγου ένωσης αφενών και ε, των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ αφετέρου είναι δύο γεγονότα που έδειξαν μια μεγάλη καμπή στην αλλαγή στις σχέσεις της Κούβας με τον κόσμο. Είναι προφανές ότι γίνονται αλλαγές γύρω από την Κούβα. Αλλαγές που δεν θέλουν είναι ταχύτερες αλλά δείχνουν ότι πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση και πρέπει να την παρακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη θα έπρεπε λοιπόν να είναι παρούσα στη διαδικασία αυτή όπως είπε ο Επίτροπος ότι γίνεται. Οι περισσότερες, ε, με τις περισσότερες χώρες ε, της Λατινικής Αμερικής έχουμε σειρά πολιτικών, οικονομικών ε, συμφωνιών. Η, Κούδα, η Κούβα είναι μία από τις λίγες εξαιρέσεις. Ελπίζω σε λίγους μήνες να υπάρχουν οι συνθήκες για να επέλθει αυτός, αυτή η συμφωνία σε πολιτικό διάλογο και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Πρόεδρε, ένα κρίσιμο κεφάλαιο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και χαίρομαι που το υπογραμμίσατε, Επίτροπε. Πριν λίγε μέρε έγινε ο πρώτος διάλογος σε υψηλό επίπεδο μεταξύ των αρχών των δύο πλευρών, Κούβας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, οι θεμελιώδει ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εσωτερικά ζητήματα, αλλά είναι βάση των αξιών τη Ένωση. Αυτή στις ε, κοινότητας ε, στις δύο πλευρές του, του Ατλαντικού, Ευρωπαίων και Αμερικανών, κοινά στοιχεία. Παρακολουθήσαμε τα δειλά βήματα της Κούβας προς τον κόσμο. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τους ίδιους τους Κουβανούς. Θέλουμε μια Κούβα που είναι πλήρως ενταγμένη στη διεθνή κοινότητα, που κερδίζει σε, σε ευημερία και σε ε, ελευθερία. Τελειώνω, η συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλά τι κάνει η Κούβα. Προσπαθεί, θέλει να συνεχίσει να διαπραγματεύεται κάτι που είναι αναγκαίο για κάθε Κουβανό. Αυτό, Πρόεδρε, θα είναι ένα επαναστατικό, πραγματικά επαναστατικό θέμα. Ευχαριστώ. Μην εκμεταλλεύεστε την ανοχή μου στο θέμα του χρόνου. Τον ε, λόγο έχει εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά ο κύριος Ζωρίνιου senhor Presidente, senhor Comissário, a União Europeia e Cuba devem. Herr Präsident, πρέπει να ε, φτιάξουμε μια ουσιαστική στρατηγική συνεργασία με την Κούβα γιατί χρειαζόμαστε εμπορικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, χρειαζόμαστε τον πολιτικό διάλογο. Πολλοί λοιπόν διαρωτούνται τι μπορεί να κάνει, ε, τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κούβα, τι μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε η Κούβα να ανοιχτεί στις ε, δημοκρατικές αξίες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε δύσκολες, ζωφερούς καιρούς, αλλά με πάση περιπτώσει παραμένει η ανθρωπιστική μας εικόνα. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι και νομίζω ότι στην Κούβα μεγάλη σημασία έχει και η κοινωνία των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε την Κούβα σε αυτό το σύστημα των εμπορικών προτιμήσεων και αυτό είναι ένα κίνητρο στην Κούβα να τηρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά κύριε Πρόεδρε, επίγει να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στην Κούβα γιατί είναι πλέον απαρχαιωμένη ε, θα έπρεπε να κρατάμε τους, ε, τις πόρτες ανοιχτές και δεν έχω κατά νου μόνο τη σχέση με την Κούβα αλλά και με τη Λατινική Αμερική και την Κεντρική Αμερική. Ο διάλογος αυτός είναι καθοριστική σημασίας ε, για βιώσιμη ανάπτυξη και λόγω της παγκοσμιοποίησης. Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών στην Κούβα και με τους θεσμούς. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις όταν πρόκειται ναι. για αξίες αλλά ε, θα πρέπει να σας πω εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών επιμένω να στηρίξουμε την ε, ύπατη εκπρόσωπο. Οφείλουμε να είμαστε ενεργοί συνεργάτες ε, στον δρόμο μιας ε, ανοιχτής δημοκρατίας, μιας πραγματικής πολιτικής συζήτησης για τις ελευθερίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή βασικών υπηρεσιών. Είναι η μόνη περιοχή στη η χώρα, μόνη χώρα στην περιοχή που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει τώρα ε, όλοι μας αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις και πρέπει να κερδίσουμε. Των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μπέλτερ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μας τους Ολλανδούς εδώ και χρόνια υπάρχουν επαφές με την Κούβα ιδιαίτερα στον θρησκευτικό θέμα. Και αυτά που μόλις άκουσα για την κατάσταση στην Κούβα σημαίνουν ότι οι επαφές με τις κουβανίδικες αρχές είναι μεν καλό πράγμα αλλά πρέπει να υπάρξουν επαφές και με τα δημοκρατικά αντιπολιτευόμενα κινήματα και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ανοίγματα στην Κούβα πράγματι και μπορεί κανείς να πει ότι οι πρωτοβουλίες της Ένωσης είναι λοιπόν θετικές αλλά χρειάζονται επαφές και για θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς στιγμήν υπάρχουν κατάφορες περιπτώσεις παραβίασης και πολιτικοί κρατούμενοι. Είναι σκανδαλώδες ότι κρατούνται πολύ όχι γιατί διέπραξαν κάποιο αδίκημα αλλά για να μην το διαπράξουν. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει επομένω κανονικές σχέσεις με την Κούβα. Για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, μετά από μήνες επιμονής ζητώντας αυτή τη συζήτηση για την Κούβα και μετά από τις πολλές καθυστερήσεις ε, συζήτησης λόγω της παρέμβασης των δύο μεγάλων ομάδων ε, του σώματος γιατί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είναι παρούσα η κυρία Μογκερίνη εδώ. Να είμαστε. Χωρίς την κυρία Μογκερίνη. Παρότι είναι παρόν ο κύριος Χάν. Είναι θλιβερό επιπλέον να βλέπουμε πως μόνο το άνοιγμα των, η αναγγελία του ανοίγματο της έναρξης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΙΠΑ και Κούβας ε, οδήγησε σε, ε, ε, σε ένα τρέξιμο των κρατών της χώρας για να εκφράσουν τη χαρά τους για την εξομάλυνση και για να φτάσουν έγκαιρα στο νησί να μοιραστούν το γλυκό. Όλα αυτά χωρίς να υπάρχουν όροι για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία χωρίς να συζητήσουν ή να συμπεριλάβουν στις συζητήσεις τους στην ε, κοινωνία των πολιτών της Κίνας, ξεχνώντας τους εκατοντάδες διαφωνούντες και αντιφωνούντες στην Κούβα που είναι χρόνια φυλακή για την πρόσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών τους. Μέσα και έξω στο νησί που, από το νησί που βλέπουν πώς ε, παραμερίζονται για την επίτευξη καλύτερων οικονομικών συμφωνιών από τις ξένες δημοκρατίες. Επιμένω εκ νέου ότι οι διαπραγματεύσει για τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας πρέπει να συνοδεύονται από μια συμφωνία χωρίς όρους για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την ανάπτυξη των ελευθεριών στο νησί. Αντίθετα, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε γι' αυτό οι ευρωπαϊκές αξίες θα πρέπει να υπερέχουν πάντα. Ευχαριστώ. Λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σοφία Σακοράφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες όπου οι ψυχροπολεμικές φωνές εντείνονται, η προσπάθεια για παραπέρα ανάπτυξη σχέσεων με την Κούβα αποτελεί απάντηση σε όσους συνεχίζουν να προτείνουν αδιέξοδες πολιτικές επεμβάσεων, αποκλεισμών και μπάρκων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μια μικρή χώρα που για πάνω από 60 χρόνια βιώνει την πίεση ενός δολοφονικού εμπάρκου προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση ισότιμα. στην πρωινή εκτενή συζήτηση για την ελλάδα αναδείχθηκε ξεκάθαρα το ουσιαστικό πρόβλημα που βιώνουν οι λαοί της ευρώπης την υποστολή και συνεχή απόσυρση του κοινωνικού κράτους και την απαξίωση θεμελιωδών κεκτημένων κάτω από την ληστρική επίθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι σε αυτή την πολιτική επιλογή αποτελεί ανάγκη να σκύψουμε με προσοχή στα όσα έχει πετύχει αυτός ο περήφανος λαός υπερασπιζόμενος την ανθρώπινη αξιοπρέπεια χωρίς να διαπραγματεύεται τις αξίες του παρά την ανηλεή επίθεση που δέχεται αυτά τα 60 χρόνια. Μια χώρα που δαπανά το 13% του αεπ της παρέχοντας καθολική δημόσια δωρεάν παιδεία με εντυπωσιακά επιστημονικά αποτελέσματα για τη διεθνή κοινότητα μια χώρα με τους καλύτερους δείκτες σε όλες τις βαθμίδες υγειονομικής περίθαλψης με δωρεάν καθολική πρόσβαση αλλά και πρωτοπόρα τόσο στον τομέα της πρόσληψης όσο και στον τομέα της διαρκούς έρευνας στο φαρμακευτικό και ιατρικό πεδίο στηρίζομαι όλες μου τις δυνάμεις στην παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεων με την κούβα με απόλυτο σεβασμό σε ένα λαό που ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες δεν εγκατέλειψε ούτε μια στιγμή την αξιοπρέπεια και το δικαίωμά του να αποφασίζει αυτός για τη ζωή του και για τη χώρα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Σακοράφα. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Χένκελ. Τη δέχεστε? Ωραία. Κύριε Χένκελ έχετε το λόγο για 30 δεύτερα. Κυρία Σακοράφα, πιστεύετε πραγματικά ότι η εξατλίωση στην Κούβα είναι η συνέπεια του εμπάργου των Ηνωμένων Πολιτειών, μα όλες οι άλλες χώρες μπορούν να έχουν εμπορικές σχέσεις με την ε, Κούβα. Θα έπρεπε ίσως ε, να μην κλείνετε τα μάτια στις αρνητικές συνέπειες του σοσιαλισμού. Εσείς τι λέτε από αυτού. Κυρία ε, Σακοράφα, έχετε τον ίδιο χρόνο για να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Χέγκελ. Κύριε Χέγκελ, δεν είναι δική μου διαπίστωση αυτή. Νομίζω ότι ολόκληρη Φίλιος αναγνωρίζει ότι επί 67 χρόνια η Κούβα στραγγαλίζεται, όπως σας θυμίζω, στραγγαλίζεται οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά και μια άλλη χώρα και μια άλλη μικρή πατρίδα, η Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίστηκαν όλα αυτά ξεπερνιούνται όλα αυτά και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άλλος δρόμος και για την ε, κούβα ένας τέτοιος δρόμος που θα την οδηγήσει ξανά στην ανάπτυξη. θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που έγινε ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που θα μπορούσε να έχει γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα απέναντι σε μια χώρα όπως είναι η κούβα. Σας ευχαριστώ κυρία Σακοράφα. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ουρτασούν. Ε, ε, Σε ευχαριστώ Δημήτρια. Είναι πάντοτε πολύ ευχάριστο να παίρνω το λόγο υπό την Προεδρία σου. Θα έπρεπε εδώ να διορθώσουμε μία ιστορική αυλεψία. Εξ ονόματος της ομάδας μου Θέλουμε να υπάρξει ομαλοποίηση των σχέσεων με την Κούβα. Τη σφερθήκαμε άσκημα το 1996 όταν δεχτήκαμε μια κοινή θέση η οποία τελικά έθεσε φρένο στη δημιουργία κανονικών σχέσεων. Γι' αυτό πρέπει να διορθωθεί αυτό το λάθος. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι ο ρόλος της Ένωσης προς την Κούβα. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο και να δώσουμε περισσότερο χώρο στην Κούβα στις ευρωπαϊκές ή στις πολυεθνικές εταιρείες. Πρέπει να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση και συνεργασία με έναν αδελφό λαό. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει γι' αυτό πολύ θετικό ρόλο. Το εμπάργκο που έπνιξε την οικονομία της Κούβας και εμπόδισε την ανάπτυξή της πρέπει απολύτως να αρθεί. Ευχαριστώ. Ελευθερίας και άμεσης δημοκρατίας ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Επιτέλους μετά από δεκαετίες υπάρχει η δυνατότητα να αρθεί το εμπάργο έναντι της Κούβας. Ένα εμπάργο που για πάρα πολλά χρόνια ε, δημιούργησε προβλήματα στον τομέα των φαρμάκων ε, στην Κούβα. Μιλάμε για μια χώρα η οποία παρά αυτές τις ε, ελλείψεις έχει το δικό μας το επίπεδο θνησιμότητας. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε το λάθος ότι να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την Κούβα. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι η Κούβα περνάει σε έναν άγριο καπιταλισμό. Ε, σήμερα ε, δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική τάξη στην Κούβα, άρα δηλαδή θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες και μεγαλύτερη φτώχεια. Το δικό μας το καθήκον είναι να στηρίξουμε τους Κουβανούς και να μην επαναλάβουμε το λάθος που κάναμε έναντι της Ρωσίας. Η συμφωνία θα πρέπει να είναι όχι μόνο εμπορική αλλά και πολιτική, να ωφελήσει τους Κουβανούς και να μην έχει ως στόχο να εκμεταλλευτούμε τις πρώτες ύλες, ε, τους ε, υδρογονάνθρακες που γίνεται για αυτούς τους λόγους σε αυτή την περιοχή. Για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας το λόγο έχει η κυρία Αρνοτή για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να χαρώ για την πρόσφατη σύναψη σχέσεων μεταξύ Ένωσης και Κούβας. Το εμπάργκο και η απομόνωση χωρών που θεωρούν μερικοί εχθρούς έχουν αποδείξει, έχει αποδειχθεί ότι δεν, δουλεύουν, δεν δουλεύει ποτέ. Δυστυχώς όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να αλλάξουν στάση μετά από δεκαετίες ενός πολύ άγριου εμπάργκο με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Κούβας. Και τελικά η Ένωση αποφάσισε στη συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτειών να συνάψει και αυτή σχέσεις. Ακόμη μία φορά λοιπόν συμπεριφέρεται σαν ουραγός και σαν υπηρέτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω οι, σχέσεις, οι καινούργιες αυτές σχέσεις να μην σημαδευτούν από το ψεύδος ο Ραούλ Κάστρο χαλάρωσε λιγάκι την αυστηρότητα του κομμουνιστικού καθεστώτος αλλά συνεχίζει να υπάρχει εδώ και πάνω από 50 χρόνια μεγάλη πολιτική καταπίεση στην Κούβα και ξέρετε ότι ο κομμουνισμός δημιούργησε παγκόσμια περίπου 100 εκατομμύρια νεκρούς. Όλοι ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά η ελπίδα αυτή δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε τι συνέβη, ότι ολόκληρες γενιές θυσιάστηκαν στο βωμό αυτής της θανατηφόρας και δικτατορικής ιδεολογίας που είναι ο κομμουνισμός. Το, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω το, τη βούληση ανοιχτών θέσεων που έχει δείξει η Ένωση έναντι της Κούβας και την προσπάθεια να υλοποιήσει μια νέα προσέγγιση για να ξεκινήσει μια πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλούμε για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Άρα πρέπει να δείχνουμε επιφυλακτικότητα όταν εξετάζουμε το θέμα της εξομάλυνσης των σιανσεών μας με αυτήν. Το, για το καθεστώς του Κάστρο, το, η θέρμανση των σχέσεων δεν σημαίνει μετά καμία διακόπτεται ο μιλητής. Η κάστα των Κάστρο με τη γερμανική διερμηνία ε, μπορείτε να με ειδοποιήσετε αν αποκαταστάθηκε είμαστε εντάξει μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Πρέντα θα το συνυπολογίσω στο χρόνο σας μπορείτε να συνεχίσετε Έλεγα για το καθεστώς Κάστρο, το, η θέρμανση των σχέσεων δεν σημαίνει πολιτική μεταρρύθμιση. Οι Κάστρο δεν έχουν καμία πρόθεση να μειώσουν τις πιέσεις προς τους πολιτικούς αντιφρονούντες. Η κυβέρνηση της χώρας συνεχίζει να ε, αποθαρρύνει κάθε μορφή κριτικής και να καταπιέζει τους αντιφρονούντες. Οι, οι, οι ειρηνικές διαδηλώσεις οδηγούν σε πανικό στο καθεστώς. Ε, πρόσφατα συνέλαβε τους, τις συζύγους των πολιτικών ε, κρατουμένων. Υπάρχουν δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι ακόμα στην Κούβα. Χιλιάδες αθώοι κρατούνται αυθαίρετα ή καταδικάζονται ενώ θεωρούν, επειδή θεωρούνται ως απειλή για το σύστημα. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης Σα θυμίζω ότι ο Γκυγέρμο Φαρίνα χρειάστηκε να περιμένει τρία χρόνια πριν λάβει το βραβείο Ζαχάροφ εδώ, γιατί οι αρχέ τη χώρα δεν του επέτρεπαν να έρθει να λάβει το βραβείο του. Η Κούβα βρίσκεται σε μια κατάσταση παρόμοια σήμερα. όποιο τολμά να ε, επικρίνει την κυβέρνηση να, να, να αναφέρει την παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου τιμωρείται αυστηρά. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την επίσημη γραμμή του κόμματο. Αυτό είναι ακριβώς η εικόνα του ολοκληρωτικού καθεστώτος. Οι εξελίξεις, οι οικονομικές αλλαγές δεν συνοδεύονται από πολιτικές εξελίξεις. Αυτό είναι μια ε, ένας, ε, μια παρακινδυνευμένη προσέγγιση. Δεν πρέπει ο καστρισμός να επανέλθει ως μια νέα μορφή αυταρχισμού όπως άλλες κομμουνιστικές χώρες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Χαουρέγγι Ατόντο. Πρόεδρε, καταρχάς να πω προς τον Επίτροπο και την ομάδα της ε, κυρίας Μογκερίνη τα συγχαρητήριά μου. Είναι σημαντικό στο σώμα να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για μια σημαντική πολιτική απόφαση της ΕΠΑ της εκπροσώπου που ήταν να πάει στην Κούβα. Η Ένωση πριν, ξεκίνησε πολλούς μήνες πριν ε, τις ΗΠΑ Πολιτείες ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με την Κούβα. Αυτό είναι σημαντικό Ήδη αυτό. Γιατί, γιατί η Κούβα είναι σημαντική. Είναι μια χώρα με μια τεράστια γεωπολιτική επίδραση στην περιοχή. Δείτε την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία για να διαπιστώσετε πόσο σημαντική είναι η Κούβα. Κοιτάξτε την ιδεολογική επίδραση που έχει η Κούβα σε όλη τη Λατινική Αμερική για να διαπιστώσετε πόσο σημαντική είναι η χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να επανέλθουν να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους γιατί θέλουν να επανέλθουν σε νέα, να επανατοποθετηθούν στη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι σημαντικό και του συγχαίρω. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην κρατάμε για την Κούβα αρχές παλιές θέσεις. Παλιέ θέσει είναι το εμπάργκο. Παλιά θέση είναι η κοινή θέση. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή θέση στι νέε συνθήκε, στου νέου καιρού που προχωρούν ταχύτατα. Δεν είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσβλέπει στην Κούβα με απλοποιημένο, απλουστευτικό τρόπο. Είτε είμαστε υπέρ είτε είμαστε κατά της Κούβας. Έτσι δεν θα λύσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την Ευρώπη που είναι να επανατοποθετηθούμε στη Λατινική Αμερική και να ανακτήσουμε ένα πολιτικό χώρο σημαντικό εκεί. Πρέπει να φύγουμε από τις απλουσευτικές προσεγγίσεις. Πρέπει να συναντηθούμε με την Κούβα. Πρέπει να υποστηρίξουμε μια δημοταβική μετάβαση, αλλά όχι απαιτώντα μια σειρά αρχών που δεν θα δεχθούν. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Η αλλαγή, η αλλαγή θα φτάσει στην Κούβα, θα φτάσει με τι εμπορικέ ανταλλαγέ, με τι προσωπικέ ανταλλαγέ, με, με το άνοιγμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθήσει η Ευρώπη σε μια μετάβαση που πρέπει να πάει προ την κατεύθυνση εκείνη. Ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γκάλερ. Τη δέχεστε. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκάλερ. Τη δέχεστε. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Είπατε ότι την αλλαγή πρέπει να τη στηρίξουμε και μέσω του εμπορίου. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν έχετε άραγε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή όσοι έχουν την εξουσία χρησιμοποιούν την απελευθέρωση στο εμπόριο για να μπορέσουν μετά από εκδημοκρατισμό να αποκτήσουν οικονομικά ωφέλη. Μήπως θα πρέπει καλύτερα να ζητήσουμε και να δούμε το θέμα καταρχήν πολιτικά. Για να απαντήσετε στην ερώτηση. Κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνουν οι αλλαγές, κανείς δεν ξέρει ε, ποιο πολιτικό σύστημα θα δημιουργηθεί εν τέλει στην Κούβα. Κατά πάσα πιθανότητα οι ανθρώπινες ανταλλαγές, οι εμπορικέ ανταλλαγές, ήδη διπλασιάστηκε ο αριθμός των Αμερικανών που έφτασαν στο νησί τους τελευταίους 6 μήνες. Διπλασιάστηκε ο αριθμός. Θέλετε με, την, ε, με τις ανταλλαγές, με το ίντερνετ, με τα μέσα επικοινωνίας, δεν πιστεύετε ότι θα φτάσει η ελευθερία, θα φτάσει. Γι' αυτό είναι έξυπνο να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε συνάδελφοι. Έστω και αν αυτοί εκμεταλλεύονται τις εμπορικές ανταλλαγές, αυτό είναι ο καλός δρόμος. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος ως εκπρόσωπος της ε, γερμανικής βιομηχανίας ε, και μακροχρόνιο μέλος της Amnesty International συναντήθηκα επανειλημμένα με τον Φιντελ Κάστρο και έχω μιλήσει μαζί του επανειλημμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τότε για την κατάργηση της ε, θρανητικής ποινή. Από το 3 ανεστάλλει, αλλά δεν καταργήθηκε. διαφωνήσαμε τότε για την κακή οικονομική κατάσταση, κακή περίθαλψη των πολιτών, σπίτια που καταραίουν στην Αβάνα και κάθε φορά έβρισκε την πρόφαση ότι αυτό οφείλεται στο αμερικανικό εμπάργο. Εγώ του είπα ότι ναι, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με την Κούβα, άρα δεν είναι αυτός ο λόγος. Όμως αυτό το αμερικανικό εμπάργο ήταν η στάνταρ πρόφασή του για να παραμείνει στην εξουσία. Κυρίες και κύριοι, αν η Αμερική τότε δεν είχε εκφράσει, δεν είχε επιβάλει το εμπάργο, οι αδελφοί Κάστρο θα είχαν εξαφανιστεί και δεν θα είχαμε και έγκλειστούς στις φυλακές. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση στην Αμερική να άρει επιτέλους αυτό το εμπάργο. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ δεν θέλω καθόλου να υπερασπιστώ τη, μια πολιτική, την πολιτική της Κούβας στις τελευταίες δεκαετίες αλλά θα ήθελα να πω ότι ο αγώνας δρόμου με τους Αμερικανούς ποιος θα είναι πιο γρήγορος για να συνάψει σχέσεις με την Κούβα ενώ δεν αλλάζουν η κατάσταση εκεί είναι και αυτός λάθος βλέπω εδώ ένα έγγραφο που υπέγραψαν χιλιάδες κουβανών για τον εκδημοκρατισμό της Κούβας έχει 10 σημεία και κανένα από αυτά δεν έχει τα αιτήματα, δεν έχει ικανοποιηθεί. Είμαι λοιπόν υπέρ μιας προσέγγισης. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να ωφεληθούμε και εμείς και οι κουβανοί, αλλά πρέπει να υπάρχουν όροι. Δηλαδή, εάν το κουβανικό καθεστώς κάνει το α θα κάνουμε το β, εάν κάνει το γ θα κάνουμε το δ. όχι υποχωρήσει μόνο εμείς και ιδίω στα δικαιώματα. Θα υπάρχουν λοιπόν όροι πρώτον και δεύτερον να απελευθερωθούν χωρίς αυτή τη φορά όρου οι κρατούμενοι. Μην αναμένετε αλλαγές σύντομα. Υπάρχουν ακόμη πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Κομισιόν λοιπόν και η Πάτη εκπρόσωπος πρέπει να δουν αυτούς τους όρους και θέλουμε αποτελέσματα. Γεια σας, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Κώστα Ντεμό. Ευχαριστώ. Τέταρτος γύρος ε, των διαπραγματεύσεων με πρόοδο. Υπάρχει πρόοδος όταν μιλάμε σε ισότιμη βάση, όταν γίνεται σεβασμός ε, του ΧΑΤΟΙΕ, της, της, της αυτοδιάθεσης των λαών. Η πέμπτο, το πέμπτος γύρος για να πετύχει το Σεπτέμβριο πρέπει να περιλάβει την κατάργηση της κοινή θέση του 1996. Είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπόδιο, πλήρες εμπόδιο στην εξομάλυνση των σχέσεων, διότι παραβιάζει την αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά ενός κράτους. Είναι και ε, πλέον ε, ε, άσχετη γιατί δεν υπάρχουν διμερείς σχέσεις. Θέλω να ζητήσω από την ΥΠΑ το εκπρόσωπη να φροντίσει, να, να παρέμβει ούτε ώστε να πάυσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε το, την, το εμπάργο και την εξοεδαφικότητα του Γκουαντάναμου. Αυτό το ζητούμε και εμείς, το ζητούν και πολλές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για την Κούβα και όχι για τη σχέση με την Κούβα. Λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρξει τάχιστα μια συμφωνία με αυτή την Ίσο οι χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ε, είναι εκείνες όπου ζει κανείς πάρα πολύ καλά. Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης, ε, της ευημερίας. Δεν ξέρω, εγώ αυτά τα αμφιβάλλω και ανησυχώ πάρα πολύ λόγω του γεγονότος ότι αυτό το άνοιγμα των Αμερικανών κατ' ουσίαν θα μπορούσε να σημαίνει ε, καπιταλιστική επιθετικότητα. Βεβαίως ε, είναι πολύ καλό το σύστημα της υγείας, της παιδείας στην Κούβα. Είναι αλήθεια ότι παραβιάζει δικαιώματα και οι πιο κατάφοροι της παραβίασης ε, είναι αυτό ε, που έκανε οι Αμερικανοί στο Κουατάνομο. Αυτό μας ενισχύει πάρα πολύ. Λέω λοιπόν εντάξει ε, καλά αυτό που γίνεται με την Κούβα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί για να μην χάνουμε τις προτεραιότητες. Ο κύριος Ούμπε Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ο σημαντικότερος εμπορικός ε, εταίρος της Κούβας ε, με κύκλο εργασιών 2 δις πέρσι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ξεκινήσει διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα και όταν πρόκειται για την ε, είσοδο σε νέες αγορές, οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωράνε ταχύτατα. Θα ήταν βέβαια καλό να ανοίξει η Κούβα. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε έξι χρόνια ε, μέχρι να δώσει κάποια εντολή. Οι Ευρωπαίοι βεβαίως έχουν ένα πολύ σημαντικό καθήκον. Ε, θα πρέπει να προβάλλουν τα καλά της Κούβας, υγεία, παιδεία και αυτά λόγω του ότι ανοίγει αγορά προς τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Έτσι λοιπόν η Κούβα χρειάζεται και μια ουσιαστική ευρωπαϊκή υποστήριξη για την οικοδόμηση ελεύθερης ε, κοινωνίας. Ελπίζω να υπάρχει μια ελεύθερη δημοκρατική Κούβα. Στα ισπανικά μιλάει ο μιλητής που συμμερίζεται τις ε, δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Επόμενος ο κύριος Βαλέζα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανοίξαμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με την Κούβα. Και το ίδιο έκαναν και οι Αμερικανοί. Αλλά οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σταθερά. Το 2015 έχουν σημειωθεί πάλι κρατήσεις αυθαίρετες. Και οι κρατούμενοι κρατούνται πολύ, πολλά χρόνια δέρνονται και δεν τους φροντίζει κανείς. Και υπάρχουν και περιορισμοί στον τύπο και στο πρόσβαση στο ίντερνετ. Οι κουβανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα σε διεθνή επιτήρηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυλακίζουν τους υπέρμαχού τους. Η Ένωση όταν έκανε τον πρώτο της υψηλού επίπεδου διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κούβα συζήτησε ζήτησε μάλλον να δημιουργηθεί ένας διάλογος επικοδομητικός και υψηλού επίπεδου αλλά δεν πρέπει να μειώσουμε τα κριτήρια μας πρέπει να ζητήσουμε πλήρη οικονομική συνεργασία αλλά που να είναι τμήμα μιας συνεχούς διαδικασίας πλουραλιστικής δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Γκίλ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, επίτροπε. Είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή που ανοίγεται προς τον κόσμο η Κούβα να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση σε σχέσεις που καλύπτουν όλα τα συμφέροντα της Ένωσης. Καλωσορίζω λοιπόν την επίσκεψη της κ. Μογκερίνης στην Κούβα τον Μάρτιο για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ε, συνεργασίας και ελπίζω να έχει την υποστήριξη των κρατών μελών για μια συμφωνία. Άκουσα με χαρά από εσά ε, την ε, έμφαση στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές ότι το εμπάργο δεν λειτουργήσε προς όφελος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ίσως ο διάλογος και η συμφωνία να αποτελέσουν ε, εργαλείο για σταδιακή αλλαγή, μια και θα επιτρέψει μια σταδιακή απελευθέρωση της Κούβας, για παράδειγμα των επικοινωνιών Πρέπει να δούμε όμως και τη γεωπολιτική παράμετρο. Η στρατηγική μας είμαι βέβαιος ότι λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις της Κούβας με χώρες όπως τη Ρωσία και την Κίνα. Η Μόσχα αποφάσισε να ανοίξει διευκολύνσεις ε, στην Κούβα ξανά και το Πεκίνο είναι βασικός εταίρος της χώρας. Τα συμφέροντα ε, αυτά συνοδεύονται και από την ε, σχέση με, την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εξετάζει αυτό η υπατή Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε θετικές εξελίξεις. Κυρίως αναφέρουμε στο ότι υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα για να υπάρχει και πολιτικός διάλογος. Εμείς βέβαια πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα στεφτεί από επιτυχία εάν ανασταλεί αυτή η πολιτική της ανάμειξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κούβα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η κουβανική κυβέρνηση τα επαναχωρήσει από το να έχουν όλοι οι Κουβανοί θέση απασχόληση. Αυτό ούτε να το φανταστούν δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Η αρχή της αυτοδιάθεσης ε, των ε, λαών με βάση των χάρτων των Εθνών πρέπει να γίνεται σεβαστή και οφείλουμε να ερωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον πιστεύει ότι θα πρέπει να χαράσετε μια πολιτική με βάση την ισότητα. Βεβαίως αυτό σε τελική ανάλυση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσύρει κανείς την άποψή του για την Κούβα. Επόμενος ομιλητής ε, για 1,5 λεπτό βλέπουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα έχουν ομαλοποιηθεί. Αυτό έχει πολλές και θετικές συνέπειες και βεβαίως ας μην ξεχνάμε αυτό θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν οι λαϊκιστές αλλά και άλλοι ακραίοι όπως ε, παραδείγματος χάρη ε, ο Μαντούρο της Βενεζουέλας. Αυτοί οι πολιτικοί ηγέτες ε, θα συναντηθούν με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ξέρουμε πως πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή την κατάσταση, να είναι μια διαδικασία για εκδημοκρατισμό σε όλη την περιοχή και όχι μόνο στην Κούβα. Για το λόγο αυτό, εγώ είμαι κατά αυτόν που λέει η Ευρωπαϊκή αριστερά, η οποία βεβαίω έχει εδώ και πολύ καιρό διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τώρα πλέον ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ανοίγουν σχέσεις με την Κούβα. Χρειαζόμαστε στρατηγικές σχέσεις ε, με τους εταίρους μας στην Λατινική Αμερική, οποτεδήποτε πρόκειται για την προάσπιση κοινών αξιών, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, πρόκειται για μια νέα Κούβα όπου δεν θα υπάρχουν πλέον πολιτικοί κρατούμενοι, όπου η ελευθερία της ε, άποψης, της γνώμης θα την χάνει εγγύησης και όπου οι κουβανοί ε, θα μπορούν να επιτρέψουν πολλά κόμματα να συμμετέχουν στις ε, εκλογές. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει στην τύχη του τον κουβανικό λαό. Η κυρία Βαλενσιάνο. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντας κάποιες παρεμβάσεις συναδέλφων, έχω την εντύπωση σαν να είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Υπάρχουν άτομα που έχουν την ίδια στάση και τις ίδιες θέσεις, παρότι στην περίπτωση της Κούβας είναι προφανής η εξέλιξη, άλλαξαν τα πράγματα. Και καθώς άλλαξαν τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωθούμε κι εμείς. Μακάρι να μην ήμασταν τόσο πίσω όσο είμαστε στη σχέση μας με την Κούβα. Πρέπει να φύγει αυτή η κοινή θέση. Το έχουμε πει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να σταματήσει το εμπάργο και να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που έγινε. Ο κ. Λαμπρινίδης ξεκίνησε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κούβα, χωρίς ωστόσο ε, να εμφανίζεται, εκεί που όμως εμφανίζεται πραγματικά ε, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σχέση με την Κούβα. Υπάρχει μια πολιτική ιστορική ναι. ανομαλία που είναι πλέον μια παθολογία σχεδόν. Πρέπει να γίνουμε πιο επίκαιροι, να αλλάξουμε την οπτική μας, να υπογράψουμε τη συμφωνία με την Κούβα και να ζητήσουμε ε, από τους Κουβανούς όπως όλους τους λαούς του κόσμου σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μακάλιστερ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κούβα αποφάσισαν ότι είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Και πρέπει οι Ευρωπαίοι νομίζω να μην παραμείνουν απλοί θεατές της αλλαγής αυτής. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή με την πρωτοβουλία του Προέδρου Ομπάμα και της κυβέρνησής του. Η σύναψη διπλωματικών σχέσεων είναι αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών καθώς και δικοματικών προσπαθειών στο Κογκρέσο. Επίσης είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών διαφόρων οργανώσεων της Κούβας. Η αλλαγή πολιτικής περιγράφεται από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μαγελθρέαος τελευταία φάση μιας πεντηκονταετούς αρνητικής εξέλιξης. Και ακόμα πιο σημαντικά πρέπει να ωφελήσει τον λαό της Κούβας πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημοκρατία στην Κούβα και με κανέναν τρόπο να μην νομιμοποιήσουμε την το αυταρχικό καθεστώς που υπάρχει εκεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι ζήτησε να συνδυαστούν οι προσπάθειες και των δύο χωρών για τη βελτίωση, αβιβαία βελτίωση και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Μιλιάν Μόν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίτροπε για τι πληροφορίε που μα δώσατε για διαπραγματεύσει τη συμφωνία με την Κούβα. Συμφωνώ, διαπιστώνω ότι προχωρούν τα πράγματα και ελπίζω η Ένωση και τα κράτη-μέλη να πετύχουν μέσω τη συμφωνία. μια σημαντικότερη και πιο ε, σημαντική παρουσία στο νησί στην κρίσιμη στιγμή που περνάει. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται μια πολιτική συμφωνία ε, και χρειά... είναι πιθανόν οι αρχές τώρα να αισθάνονται λιγότερο αναγκασμένες να έχουν μια συμφωνία με την Ευρώπη μετά την εξομάλυνση των σχέσεών τους με τη, με τη ΣΥΠΑ. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πέραν κάποιων μικρών αλλαγών ε, δεν άλλαξε ριζικά η φύση του καθεστώτος την Κούβα. Τον Ιούνιο έγινε μια πρώτη συνάντηση για ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ του κ. Λαμπρινίδη, ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ένωσης και των υπευθύνων της Κούβας. Εμείς επιμείναμε στο ζήτημα αυτό, ζητώντα να αλλάξει για παράδειγμα η ποινική νομοθεσία της, να επικυρώσει τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και για τα κοινωνικά δικαιώματα που έχει μόνο υπογράψει. Mm. Όπως γνωρίζετε δυστυχώς συνεχίζονται οι αυθαίρετες πράξεις, η παρενόχληση των ε, υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σας παραπέμπω στην έκθεση, την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου και τα λόγια που μας είπε ο κ. Χάν όταν μας ενημέρωνε την περασμένη εβδομάδα. Κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Αμερική συνδέονται με μια σειρά αξιών mm προστασία του κρατου δικαίου, τη δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κούβα δεν μπορεί να είναι εξαίρεση. Εγώ ελπίζω να συνεχιστούν οι συναντήσει που ξεκίνησαν στις 25 του μηνό Ιουνίου και να υπάρξει μια ε, πραγματικά προ, των σχέσεών μας. 1,5 λεπτό κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ πιστεύω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε μια επικοδομητική πολιτική έναντι της Κούβας και πρέπει να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων στην Κούβα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από τη μετάβαση ε, κομμουνιστικών καθεστώτων σε δημοκρατικές κοινωνίες και νομίζω ότι οι Κουβανοί θέλουν τον εκδημοκρατισμό. Δεν πρόκειται ε, για συνέχιση κομμουνιστικής ε, δικτατορίας ούτε για κονκίστα από το Μαϊάμι. Κάπου στη μέση θέλουν να κινηθούν οι άνθρωποι και νομίζω ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να σφυριλατήσουν μια κουβανική κοινωνία που θα είναι γνήσια, κουβανική η Κούβα δεν έχει απαραίτητα ε, κομμουνιστικό ε, καθεστώς, ε, ούτε και το Μπατίστα βέβαια ένα τέτοιο κόμμα, το αυτό πρέπει να επαναφέρει κανείς. Ε, η δημοκρατία υπάρχει σε πάρα πολλές μεταβατικές κοινωνίες. Όπως και ο συνάδελφος Χένκελ και εγώ πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχουν άρει το εμπάργο, όπως έγινε και με το τείχος του Βερολίνου. Και αν γινόταν αυτό δεν θα είχε φτάσει η χώρα εκεί που έφτασε σήμερα, θα είχε υπάρξει εκδημοκρατισμός πολύ νωρίτερα. Έτσι λοιπόν ε, με τις ε, ε, προσφορές που κάνουμε να θέσουμε και προαπαιτούμενα με στόχο η δημοκρατική αντιπολίτευση στην Κούβα να έχει προοπτική μέλλοντος, να τα διαπραγματευτούμε αυτά με το καθεστώς, το πότε θα είναι οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές στην Κούβα, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Διαδικασία του Κατσιάη τώρα. Επτά αγορητές. Πόλτσακ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχήν, οτιδήποτε έζησε τα τελευταία δεκαετίες η Κούβα είναι φοβερό βάρος και θα ήταν σωστό να ελαφρυνθεί αυτό. Η Ένωση έχει ήδη αρχίσει αλλά νομίζω ότι πρέπει να τεθούν όροι, πρέπει να θέσουμε όρια και να προστατέψουμε τουλάχιστον τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό συνυπογράφω την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δόγμα του Βάτσλαβ Χάβελ, πρώην Προέδρου μας, ότι θεωρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασική αρχή αναφέρετη που δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με κάτι χαμηλότερης αξίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διαπαρατευόμαστε προς το συμφέρον του κουβανικού λαού αλλά να υπάρξουν όρια και όρια. Ευχαριστώ. Ποιος? Φρουντσούλικα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει μια νέα περίοδο σχέσεων μεταξύ Ένωσης και Κούβας βάσει της ανάγκης να προωθήσουμε την δημοκρατία στη χώρα και την ενθάρρυνση οικονομικών αλλαγών. Πρέπει να συνοδεύσουμε την Κούβα στην συνεχιζόμενη διαδικασία εξυγχρονισμού και να προωθήσουμε την, τον πολιτικό διάλογο για ζητήματα όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ελευθερία έκφρασης αυτή τη σημαντική διαδικασία εξέλιξης. Η Κούβα μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας των χωρών ΑΚΕ, υποστηρίζοντας το αίτημα αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Κούβας και δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ με στενή συνεργασία και βελτιώνοντας τις σχέσεις. Και οι δύο πλευρές θα κερδίσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει για ένα λεπτό. Των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για την Ένωση στο σύγχρονο πολυπολικό κόσμο που ζούμε στο πλαίσιο αυτό η αποκατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Κούβα αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώ η ένωση μέσω τη εξωτερική τη πολιτική θα μπορούσε να αποκτήσει μια ανεξάρτητη θέση έναντι αυτής των ηνωμένων πολιτειών τη Αμερική. Βεβαίω η αποκατάσταση των σχέσεων ηπα κούβας οπωσδήποτε θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων τη Κούβα με τον δυτικό κόσμο. θεωρούμε σημαντικό το διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση Κούβα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για έμεση επέμβαση της ευρωπαϊκής ένωσης στα εσωτερικά της κούβας. θεωρούμε σημαντική τη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων ευρωπαϊκής ένωσης κούβας προσέγγιση όμως που θα πρέπει να γίνει στη βάση της αρχής του αμοιβαίου ωφέλους και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. τέλος η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να πάψει να εποφθαλμιά την εκμετάλλευση των πλούτοπαραγωγικών πηγών της κούβας αντί πινακίου φακής. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με ανθρώπους ε, στην Κούβα που είναι στη φυλακή, ε, με ψεύτικες κατηγορίες. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με ανθρώπους στη Βαρκελόνη. Και έτσι λοιπόν ένιωσα την ελπίδα τους πολλές προσδοκίες ε, που εκφράζονται έναντι ημών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν και επιθυμούν τη δημοκρατία ε, πρέπει να στηριχθούν από εμάς. Ε, στηρίζω την ομαλοποίηση και με τον νυν καθεστώς. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόοδος ε, προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Βεβαίως και βοηθούν οι οικονομικές σχέσεις, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λαός υποφέρει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλουμε να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην νήσο, στο κουβί, στην Κούβα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για όλους για τη συζήτηση συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούστηκαν όλοι να λένε ότι το εμπάργκο δεν έχει λύσει τίποτα η υπογραφή ανούσιων συμφωνιών δεν έχει κανένα, κανένα αποτέλεσμα. Αυτά είναι πράγματα του παρελθόντος. Αν θέλουμε να αρχίσουμε μία αληθινή εταιρική σχέση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και εμείς έχουμε κάνει πολλά λάθη στην εξωτερική μας πολιτική στο παρελθόν και πρέπει να αρχίσουμε να τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα, για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε μία δουλειά, σε κάποια εκπαίδευση Όλα αυτά είναι κανονικά ανθρώπινα δικαιώματα που εφαρμόζονται και στην Κούβα. Είναι όμως κανονικά ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρώπη. Πρώτα να, να καθαρίσουμε τα του οίκου μας και μετά να κατηγορήσουμε την Κούβα. Να δούμε πώς ζουν στην Κούβα οι άνθρωποι και πώς ζουν στην Ευρώπη. Είμαι ευγνώμων στην υπάτη εκπρόσωπο για ό,τι έκανε και νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να συνάψει σοβαρή σχέση με την Κούβα. Σας ευχαριστώ. Ο Σόλτ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, για πολλά χρόνια η Κούβα ήταν ένα θέμα ταμπού. Για πολλά χρόνια ήταν μια χώρα απομονωμένη από την οικονομική συνεργασία και με την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είχε επιπτώσεις, συνέπειες και στις δύο πλευρές. Καλωσορίζω λοιπόν τις ε, προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων με την Κούβα και για την υπογραφή μιας συμφωνίας με τη χώρα. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις προσπάθειές μας αυτές. Πρόκειται για μια χώρα που δεν μας επιτρέπει να επιβάλλουμε την δημοκρατία μας σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται την ποικιλομορφία τη διαφορετικότητα και να αναγνωρίσει το δικαίωμα των λαών της Κούβας να αποφασίσουν για τον εαυτό τους. Αν δούμε, αν διαβάσουμε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ εδώ στο Στρασβούργο, βλέπω ότι μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα απαντήσει κλείνοντας ο κύριος Χάν μιλώντας εξ ονόματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ ευχαριστώντας για αυτή τη συζήτηση και πάλι και για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ Κούβας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο από πλευράς ε, Μπαραντιάραν που αναφέρθηκε πιο πριν ότι δεν, δεν είναι παρούσα η κυρία Μογκερίνη και εξέφρασε την ε, δυσφορία γι' αυτό και ο λόγος για την απουσία της είναι απλώς Συμμετέχει στις ε, διαπραγματεύσεις στη Βιέννη μεταξύ των δυνάμεων και του Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό είναι επαρκής δικαιολογία για την επίτευξη σε συμφωνία το δυνατόν ταχύτερα. Και επανέρχομαι στη συζήτηση ήθιστε σε τέτοια θέματα οι συζητήσει να αντανακλούν ένα ευρύτερο, ε, μεγάλο εύρο θέσεων που δεν είναι πάντα εύκολο να συγκλίνουν. Έχοντας παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν, αισθάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη σωστή οδό, στη σωστή πορεία με την κατεύθυνση που υιοθετήθηκε το 2014. Μια πιο στενή σχέση συνεργασίας με την Κούβα ώστε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και να βρούμε ειρηνικούς τρόπους ε, για να προωθήσουμε αμοιβαία συμφέροντα. Η συμφωνία συνεργασίας ε, θα είναι ένα σημαντικό βήμα ακριβώ προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έδινε μια ικανή πλατφόρμα για έναν ικανό επικοδομητικό διάλογο και χρηματοοικονομική συνεργασία και παγίωση της συνεργασίας και δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης που είναι θεμελιώδη θέματα ώστε να μπορέσει αυτή η σχέση μας να αναπτυχθεί παράλληλα με τις αξίες μας. Και το βίωμα αυτό, η εμπειρία αυτή θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για τον κοινωνικό εξυγχρονισμό μπορεί να δείξει, να καταδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μια οικονομία της αγοράς μπορεί να συνδυάζεται με υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και ταυτόχρονα συμμετοχή των πολιτών. Πολλοί από εσά εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εκ του σύνεγγυς πολύ προσεκτικά παρακολουθούμε αυτά τα θέματα και τις ανησυχίες που όπως εξεφράστησαν ήδη στην εισαγωγική μου παρέμβαση είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό το θέμα το θίγουμε σε τακτά διαστήματα συστηματικά με τους κουβανούς εταίρους μας και έχουμε ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις ήδη πριν από την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια βάση για επικοδομητικές συζητήσεις το δυνατόν νωρίτερα. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέρος της ιστορικής διαδικασίας που τεκταίνεται αυτή τη στιγμή στην Κούβα, <clears throat> θα πρέπει να στοχεύει στο να μπορέσει να προωθήσει αυτή τη διαδικασία, να ενθαρρύνει τι μεταρρυθμίσει και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ένα πράγμα λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να εμπλακούμε σε αυτές τις διαδικασίες με την Κούβα. Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε και στο μέλλον. La discussione sulle... Η συζήτηση όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής